Κυρίες και κύριοι, κύριοι, ε, αγαπητοί συνάδελφοι, ας ε, ξεκινήσουμε την απογευματινή συνεδρίαση όπου έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε και καταρχήν ε, θεωρώ ότι έχουμε αρκετούς παρισταμένους. Καταρχήν έρχομαι στο σημείο 7, κατάρτιση μιας νέας Ευρωπαϊκής Ατζέντας για την Ψηφιακή Τεχνολογία 2015 και η συγγήτρια είναι η Πιλάρ Δεκαστήλινο που έχει το λόγο. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, ε, βρισκόμαστε στην τελευταία συζήτηση, η οποία θα εστιάσει κυρίως ε, στις τροπολογίες για τη νέα ε, ψηφιακή ατζέντα 2015.eu η κατάσταση μέχρι του έχει ως εξής. Δεν ε, προβλέπονται αλλαγές. Καταρχήν ε, υπάρχει συμφωνία και πρέπει να πω ότι μιλάμε για συμφωνία για όλες τις πολιτικές ομάδες ε, της Επιτροπής μας. Ε, έχουμε 28 τροπολογίες ε, συμβεβαστικές και σε αυτές τις τροπολογίες καταλήξαμε, προσπαθήσαμε να καταλήξουμε σε μια συμβεβαστική θέση, σε μια κοινή θέση για αυτή την ψηφιακή ατζέντα. Ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις πολιτικές ομάδες, όλους τους σκιώδεις συγητές από όλες τις πολιτικές ομάδες και τις προσπάθειες που έκαναν ώστε να μπορέσουμε αύριο να έχουμε αίσιο αποτέλεσμα. Ε, πριν πω λοιπόν οτιδήποτε άλλο να τους ευχαριστήσω. Το τελικό αποτέλεσμα που θα είναι και η θέση του Κοινοβουλίου που θα εκφραστεί αύριο στην Επιτροπή Ήτρε και κατόπιν τον επόμενο μήνα θα είναι η θέση στην Ολομέλεια. Ελπίζω να έχουμε μια θέση αντίστοιχη με αυτήν που θα επιτύχουμε αύριο εδώ. Και μιλάμε για μια θέση η οποία είναι καταρχάς πολύ επίκαιρη, διότι βρισκόμαστε σε μια χρονική συγκυρία στην οποία όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα από το Συμβούλιο μέχρι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Προεδρία αυτή τη στιγμή, την Ισπανική Προεδρία, αναπτύσσουν προτάσεις προς την ίδια κατεύθυνση με τον ίδιο στόχο. Ο στόχος είναι να έχουμε ένα στρατηγικό πλαίσιο προσανατολισμού προκειμένου να δημιουργήσουμε τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να εκμεταλλευτεί στο μέγιστο όλες τις δυνατότητες που προσφέρει αυτή η, ψυχιακή, η ψηφιακή εποχή, ε, αυτή η ε, ψηφιακή πλατφόρμα, αν μπορούμε να την αποκαλέσουμε έτσι. Το Κοινοβούλιο έχει πλέον μια πρώτη θέση, η οποία νομίζω ότι θα πρέπει να μας ικανοποιεί. Είναι μια θέση η οποία προέκυψε από πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, νομίζω τον Αύγουστο, ε, ζήτησε μία αξιολόγηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το Κοινοβούλιο για το τι ακριβώς θα έχουμε το 2010. Το Κοινοβούλιο ανέλαβε την πρωτοβουλία να κάνει μία έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας και αυτό θα έχουμε αύριο, θα έχουμε μία ψηφοφορία που θα δώσει ουσία σε αυτή τη θέση του Κοινοβουλίου. Το πακέτο τηλεπικοινωνιών βλέπει το φως ε, και ταυτόχρονα έχουμε υποστήριξη ε, και από το Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, όλα τα θεσμικά όργανα οδεύουν προς την ίδια κατεύθυνση. Θέλουμε να έχουμε ευνοϊκές συνθήκες για να έχουμε επενδύσεις, να υπάρχει βεβαιότητα για το εμπόριο, να υπάρχει προστασία των καταναλωτών και πολλά άλλα πράγματα. Και το επόμενο βήμα ή μάλλον για να το πω καλύτερα, τα επόμενα βήματα είναι δύο. Να έχουμε ε, ταχεία, συνεκτική και συνεπή εφαρμογή του πακέτου των τηλεπικοινωνιών σε όλα τα κράτη-μέλη, γεγονός που αποτελεί ικανή και αναγκαία συνθέκη, προκειμένου στη συνέχεια η ψηφιακή ατζέντα και όλα όσα περιέχει η ψηφιακή ατζέντα και θα περιέχουν οι ψηφιακές ατζέντες σε εθνικό επίπεδο να μπορέσουν να αναπτυχθούν. Και για να γίνει κάτι τέτοιο δεν έπρεπε να περιμένουμε μέχρι να εφαρμοστεί το πακέτο των τηλεπικοινωνιών, αλλά να έχουμε ένα πλαίσιο ε, στρατηγικής αναφοράς, το οποίο θα μας δώσει κάποιους προσανατολισμούς για τομείς δράσης, για συγκεκριμένους στόχους και για συγκεκριμένους ε, πτυχές τις οποίες μπορούμε να αναπτύξουμε για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Αυτό ακριβώς είναι η ψηφιακή ατζέντα είναι ένα πλαίσιο αναφοράς, στρατηγικής αναφοράς, το οποίο συμμερίζονται όλοι και έχει ένα πολύ συγκεκριμένο περιεχόμενο, αναφέρεται σε συγκεκριμένους τομείς δράσης, με συγκεκριμένους στόχους και μέσα τα οποία επιτρέπουν να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Δεν θα επισέλθω εκ νέου σε λεπτομέρειες, διότι νομίζω ότι δεν είναι απαραίτητο, δεν χρειάζεται να εξηγήσω από την πλευρά του Κοινοβουλίου ποια είναι τα βασικά θεμέλια πάνω στα οποία έχει οικοδομηθεί αυτό το πλαίσιο στρατηγικής αναφοράς. Ωστόσο, δεν θα ήθελα να μην αναφέρω δύο πολύ σημαντικά στοιχεία. Πρώτον, το επίκεντρο για όλη αυτή τη δράση, για όλες αυτές τις ε, ε, δράσεις, αυτό το πλαίσιο αναφοράς στην ψυχιακή εποχή είναι ο άνθρωπος, ως καταναλωτής και ως πολίτης. Και επομένως, η, η ενδυνάμωση και η διευκόλυνση των ανθρώπων προσφέρονται τους τα κατάλληλα μέσα. Το να διευκολύνουμε τους ανθρώπους με το ε, να τους προσφέρουμε τα δίκτυα τα οποία θα τους επιτρέψουν να λάβουν τις πληροφορίες, τις ευκαιρίες, ε, με όλες τις έννοιες και την ε, διασφάλιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών στο ψηφιακό πεδίο είναι κάτι το οποίο είναι θεμελιώδες. Σε αυτό λοιπόν το σπήρωμα το οποίο παρουσιάζεται μέσα σε αυτή την ε, πρόταση, ο άνθρωπος είναι στο κέντρο αυτού του ελατηρίου, αυτού του σπηρώματος. Και θα ήθελα να σταθώ και σε ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο θεωρώ πολύ ουσιαστικό. Η ψηφιακή ευρωπαϊκή ενιαία αγορά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε ακόμα ενιαία αγορά, μόνο ένα 7% έχουμε βαρεθεί να το επαναλαμβάνουμε αυτό, μόνο ένα 7% των συναλλογών που γίνονται στο διαδίκτυο από πλευρά Ευρωπαίων καταναλωτών είναι διαμεθοριακές. Ενώ όλε οι υπόλοιπε συναλλαγέ γίνονται ε, εντός των κρατών μελών. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένας τεράστιος κατακαιρματισμός της αγοράς, ε, ο οποίος αποτελεί πρόσκομα, διότι δεν μπορούμε έτσι να αναπτύξουμε όλες αυτές τις δυνατότητες που έχουν να προσφέρουν τα 500 εκατομμύρια καταναλωτών σε ένα χώριο όπως είναι το διαδίκτυο στην ψηφιακή εποχή. Θα πρέπει λοιπόν να αρθούν τα νομικά εμπόδια τα οποία δεν επιτρέπουν την εξέλιξη αυτής της ενιαίας αγοράς, η οποία αγορά θα πρέπει να είναι ανοιχτή και ανταγωνιστική τα επίπεδα ανταγωνισμού αυτής της αγοράς είναι καθοριστική σημασίας Κατά πρώτον, διότι θα υπάρχουν δυνατότητες για τον κάθε έναν από εμά. Υπάρχουν περισσότερες εναλλακτικέ λύσεις και θα υπάρχουν ταυτόχρονα και ανταγωνιστικές τιμές, οι οποίες ε, είναι πολύ σημαντικές, ώστε να μπορούν οι άνθρωποι από εκεί και πέρα να αποκτούν όσο το δυνατόν περισσότερα πλεονεκτήματα. Συνοψίζοντας, κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, δεν θα ε, μακρηγορήσω άλλο. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα χρονική στιγμή, η οποία συμπίπτει και με την έναρξη της θητείας μας, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα και στους ευρωβουλευτές μέλη αυτού του Κοινοβουλίου ένα χρονικό ορίζοντα άνω των τεσσάρων ετών για να μπορέσουν να συνεχίσουν να οθούν μέσω της αξιολόγησης και της εποπτείας ε, το θέμα αυτό. Γι' αυτό λοιπόν ζητάμε να υπάρχει και ένας πίνακας αποτελεσμάτων, ένα scoreboard, το οποίο θα μας δίνει τη δυνατότητα ε, να παρακολουθούμε μία σειρά από ευρωπαϊκούς και εθνικούς στόχους. Ε, υπάρχει το ετήσιο ε, γιατί η ετήσια σύνοδος ε, ψηφιακών θεμάτων, το Annual Digital Summit, το οποίο θα συζητά όλα αυτά τα θέματα και την εξέλιξη αυτού του ε, τεράστιου αμαλγάματο ε, θεμάτων και ευκαιριών που προσφέρονται από την ψηφιακή επανάσταση. Τίποτα άλλο και ευχαριστώ πολύ εκ νέου σε όλου. Ευχαριστώ. Η κυρία Βάλιαν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ε, συγχαρώ την εισηγήτρια για την εργασία και για την πρόοδο που έδειξε. Υπάρχουν ορισμένες τροπολογίες τις οποίες καταθέσαμε με πάρα πολύ μικρή προθεσμία. Είναι σημαντικό να δούμε το θέμα των συμβιβαστικών τροπολογιών που θα το δούμε αύριο ε, για να στείλουμε ένα πολύ σαφές και πακριβές μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, με ανησυχεί, δεν ανησυχώ για την τύχη της έκθεσης, αλλά με ανησυχεί η στρατηγική, αν θέλετε, ε, την οποία προβλέπουμε. Δεν θέλουμε να γίνει ένα πεδίο πάρα πολύ ευρύ που κυνηγάει πάρα πολλούς στόχους και παραμένει ασαφές. Γι' αυτό οι συμβαστικές τροπολογίες κατά την άποψή μου δίνουν μια πολύ καλύτερη στόχευση από αυτές που κατατέθηκαν. Ε, πρέπει να γίνει μια ε, αναπροσαρμογή της ε, στάσης των ενιαίων υπηρεσιών για την τροπολογία 5 το να μην υπάρξει επιπρόσθετος φόρτος στου καταναλωτές και τους χειριστές. Αυτό είναι μια τροπολογία η οποία αφορά το ταμείο που θα ασχοληθεί για αυτόν τον στόχο και η οποία θα πρέπει να προσέχει να μην γίνεται διαστρέβλωση του ανταγωνισμού λόγω των εξωτερικών επενδύσεων. Ύστερα χαιρετίζω το γεγονός ότι εκτός του ότι οι πολίτες βρίσκονται σε μια κατάσταση που τους αφαιρείται η κάθε αρμοδιότητα και εξουσία μέσα στην κοινωνία με τη συμβαστική τροπολογία ε, γίνεται, προτείνεται ένας ανταγωνισμός μεταξύ των δύο δομών και ε, του, της Telecom και των ανταγωνιστών της για να προωθηθούν οι επιχειρήσεις και οι Επίσης χαιρετίζω την, την αλλαγή του περιεχομένου, την εξέλιξη ε, στον βιομηχανικό τομέα, όπου τονίζεται όχι μόνο η εξέλιξη της ε, συμπεριφοράς ως προς το ε, το, το καινούριο περιεχόμενο. Υπάρχει το θέμα της στήριξης του καινούριου περιεχομένου από τη μία πλευρά και από την άλλη τη στήριξης των όσων έχουν πνευματικά δικαιώματα. Δεν γίνεται ωστόσο κανένα ε, καμιά αναφορά στο περιεχόμενο και στις σχετικές βιομηχανίες. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να ε, μπούμε, να επισέλθουμε μέσα στο χώρο το, της πνευματικής ιδιοκτησίας όπου οι διακρίσεις είναι πάρα πολύ λεπτές και τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Ο Ιταλός ε, συντονιστής ε, μας ικανοποίησε πάρα πολύ σε ό,τι αφορά το σπέκτρουμ και ε, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να περιορίσουμε αυτές τις αρμοδιότητες για να έχουμε ένα καινούριο σπέκτρουμ που να μην βλάπτει τις δραστηριότητες στις χώρες μέλη. Επίσης το αίτημα για ίντερνετ και για τις υπηρεσίες IT ε, είναι προσπάθειες που έχουν εστιαστεί σε ορισμένα μέτρα που λαμβάνονται για τη σωστή παροχή και κάλυψη των δικτύων και για τα δίκτυα υποδομών. Αυτά τα μέτρα είναι πάρα πολύ σημαντικά οπωσδήποτε και πιστεύουμε ότι πρέπει να συγκεντρωθούμε, ε, να επικεντρωθούμε σε αυτά. Ε, το broadband internet επίσης το είναι πάρα πολύ σημαντικό και το ευρυζωνικό διαδίκτυο ε, πρέπει να προωθηθεί. Υπάρχει ο σχετικός κανονισμός ε, ο οποίος εκπονείται. Ε, υπάρχουν εταιρείες οι οποίες δεν μπορούν να κατανοήσουν το πώς, θα χρησιμοποιηθούν, το πώς οι χρήστες θα δρουν μέσα σε αυτά τα καινούργια δεδομένα. Γι' αυτό όλα αυτά πρέπει να γίνουν πιο στο μέτρο του δυνατού και θα πρέπει να βρούμε και την νεότερη, την τελευταία εκδοχή γιατί αυτή που προτάθηκε δεν ήταν ε, ικανοποιητική. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κύριος Κάλφιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα κι εγώ να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή, την ε, κυρία Δελκαστίγιο για την εργασία που έχει κάνει σε αυτό το θέμα και για την εξαιρετική συνεργασία την οποία ε, είχαμε κατά την διαμόρφωση του κειμένου που θα προταθεί. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από πολλούς ενδιαφερομένους στα κράτη-μέλη σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ε, ε, για διατύπωση τροπολογιών και νομίζω ότι μία τη πρόταση του, της συγγήτριας ήταν να επικεντρώσουμε τη συζήτηση βρίσκοντας τα θέματα τα οποία πρέπει να προχωρήσουν στο διάλογο προτού δημοσιεύσει την ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά είναι μια εξαιρετική πρόταση για να μην επαναφέρουμε θέματα τα οποία έχουν ήδη συζητηθεί και εκ των οποίων έχουμε δει διάφορες μορφές όπως στο θέμα των τηλεπικοινωνιών και ούτω καθεξής. Άρα να μην ξαναανοίξουμε το θέμα αυτό, να ζητήσουμε μία εφαρμογή, να πάμε ένα βήμα παραπέρα και νομίζω ήταν πολύ καλή λύση. Η ιδέα της εκθέσεως είναι να δώσει ένα πολύ ευρύ πολιτικό μήνυμα εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στη συνέχεια να αναμείνει την ανακοίνωση του, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα κοινοποιηθεί στο τέλος του επομένου μηνός και να συζητήσουμε τα θέματα αυτά όσο το δυνατόν πιο ειλικρινά. Βεβαίως είχαμε διάφορα σημαντικά θέματα σαν σοσιαλιστές και δημοκράτες ε, για την εργασία σχετικά με αυτό το θέμα. Θα αναφερθώ σε λίγα από αυτά. Ε, βεβαίως ε, ήμασταν πολύ θετικοί και προσπαθήσαμε να βρούμε ε, ως το δυνατόν περισσότερη όθηση για, ε, για επενδύσεις και για ανάπτυξη του διαδικτύου. Συγχρόνως όμως θα πρέπει να γίνει και μία ψηφιακή αλλαγή και θα πρέπει να σκεφτούμε τους καταναλωτές οι οποίοι να έχουν δυνατότητα πρόσβασης ε, σε μία αποδεκτή, σε ένα αποδεκτό κόστος. Δεν πρέπει δηλαδή να προωθηθεί το θέμα αυτό μόνο προς όφελος των επιχειρήσεων και των βιομηχανιών αλλά και ε, σε ε, όλους τους τομείς της δημοσίας ζωής και είναι πολύ σημαντικό πλέον το διαδίκτυο για τους καταναλωτές και ιδίω για αυτούς οι οποίοι ε, είναι στο περιθώριο και δεν λαμβάνονται πάντοτε υπόψη διότι ζουν σε απόμακρες περιοχές, ότι δεν έχουν σταθερή απασχόληση και πολλές φορές όλα αυτά τα άτομα δεν τα λαμβάνουμε υπόψη όταν σκεφτόμαστε νέες γενναίες για την παροχή υπηρεσιών. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν θα πρέπει το θέμα αυτό να μας απασχολήσει ιδιαιτέρως. Όπως και για πολλούς συναδέλφους από άλλες ομάδες ήταν πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την ουδετερότητα. Μία αρχή η οποία ε, είναι πολύ σημαντική και πρέπει να διατηρηθεί εάν θέλουμε παρκή χώρο για να ε, υποκινήσουμε περαιτέρω εξέλιξη του διαδικτύου. Συγχρόνως υπάρχει ο ρόλος των ε, ε, μέσων αυτών για να ενισχύσουν την οικονομία και να ανοίξουν δυνατότητες για το κοινό. Αυτό που μας απασχολεί είναι τα θέματα που έχουν σχέση με την ασφάλεια και ε, δεν είναι το σημείο όπου θα λύσουμε όλα τα θέματα διότι ξέρω ότι και οι νομικές υποθέσεις, η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων ασχολείται με ε, την ε, με ε, ε, τις νομικές πτυχές και ε, γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι πολύ βασικό να μπορέσουμε να εστιαστούμε στα θέματα τουλάχιστον για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες διότι θα μπορέσουμε νομίζω να καταλήξουμε σε έναν αποδεκτό συμβιβασμό αποδεκτό τουλάχιστον για όλες τις μεγάλες πολιτικές ομάδες και συγχρόνως να δώσουμε ένα ηχηρό μήνυμα από πλευράς του Κοινοβουλίου για την εξέλιξη αυτών των θεμάτων. Οι συμβιβαστικές τροπολογίες έχουν ε, καλέψει ε, τα περισσότερα θέματα και ε, τη χάνουν τη συνένεση σχεδόν όλων των πολιτικών ομάδων. Δεν θα ήθελα εδώ να αναφερθώ σε όλα τα σημεία που μας χώριζαν και γι' αυτό επιλέξαμε να δώσουμε ένα ηχηρό μήνυμα πολιτικό για το πόσο μας ενδιαφέρουν αυτά τα θέματα. Υπάρχουν βέβαια λεπτομέρειες οι οποίες πρέπει ακόμη να τελειοποιηθούν και ελπίζω ότι θα είναι μια πολύ αποτελεσματική απόφαση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Έντσου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ την κυρία Καστίγιο για την προσπάθεια που έκανε να συντάξει αυτή την έκθεση. Σίγουρα δεν ήταν δύσκολο, εύκολο συγγνώμη, το έργο της. και εκτιμώ και τη συνεισφορά των συναδέλφων υπομορφή τροπολογιών. Η ψηφιακή ατζέτα και μια ενιαία αγορά πληροφορικής ε, είναι μία από τις προτεραιότητές μας, μία προτεραιότητα άλλωστε και της Προεδρίας. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τον 21ο αιώνα χωρίς να σκεφτόμαστε το διαδίκτυο, τα δίκτυα επικοινωνίας και ούτω καθεξής. Χαιρετίζω το γεγονός λοιπόν ότι σε αυτή την έκθεση εστιάζουμε στην ε, ολοένα αυξανόμενη ε, ψηφιακή γνώση που αποκτούν οι νέοι άνθρωποι, διότι είναι αυτοί που χρησιμοποιούν περισσότερο τις νέες τεχνολογίες. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ασφάλεια και αποτελεσματικότητα στην χρήση του διαδικτύου. Επίσης, θα πρέπει να υπάρξει ίσως και μια εκστρατεία η οποία θα φορά ενηλίκους και κυρίως γονείς και θα τους βοηθήσει να εκπαιδεύσουν και να προστατεύσουν τα παιδιά τους ε, τα οποία θα ζουν σε ένα ψηφιακό κόσμο ε, και να προστατεύεται αφενός η ιδιωτική τους ζωή αλλά και η ασφάλειά τους. Κάτι ακόμα το οποίο θα ήθελα να επισημάνω είναι το θέμα της οικονομικής ε, προόδου, της ανεργίας και των οικονομικών προβλημάτων. Ε, η τροπολογία 166 ζητά από, τα κράτη, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συντάξει ένα πρόγραμμα για να προαγάγει τις ε, επιχειρήσεις online και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας για ανθρώπους που έχασαν πρόσφατα τη δουλειά τους. Θα ήθελα να ζητήσω λοιπόν την υποστήριξή σας για την τροπολογία αυτή και ταυτόχρονα θα ήθελα να ζητήσω και την υποστήριξή σας εκ μέρους των Ευρωπαίων πολιτών. Θα πρέπει να τους δώσουμε μια νέα ευκαιρία. Μέσω τέτοιων εργαλείων θα μπορέσουμε να μειώσουμε ουσιαστικά τον αριθμό των ανέργων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό συμπεριλαμβάνεται μεν στη συμβιβαστική τροπολογία, αλλά δεν καλύπτει την κοινωνική πτυχή της πρότασής μου. Ε, θα πει κανείς ότι τα κοινωνικά θέματα δεν είναι θέμα ε, αυτής της έκθεσης, αλλά οι Ευρωπαίοι πολίτες ε, στρέφονται σε εμά ε, στα μέλη της Επιτροπής ε, Ήτρε και ψάχνουν μία ένδειξη υποστήριξης σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς. Ευχαριστώ, η Αγγέλη Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εξαιρετική εργασία της. Η κυρία Καστήλιο όχι μόνο κατήρθησε μια εξαιρετική έκθεση, αλλά όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, κατάφερε πάρα πολύ γρήγορα να οδηγήσει τις πολλαπλές τροπολογίες σε συμβιβαστικές, οι οποίες θα υπερψηφιστούν πιο εύκολα. Την ευχαριστώ και νομίζω ότι είναι μια καλή αρχή εδώ στην Επιτροπή μας επί του θέματος. Υπάρχουν δύο θέματα τα οποία θέλω να θίξω και στα οποία έχουν αναφερθεί οι συνάδελφοι. Νομίζω ότι κατόπιν των τελευταίων πέντε ετών ή τουλάχιστον των ετών από όταν συζητάμε τα θέματα των τηλεπικοινωνιών ή στο Κοινοβούλιο να έχουμε αποκρισταλώσει κάποια γνώμη. Άρα τώρα πρόκειται ε, για την εφαρμογή ε, των συμβιβαστικών λύσεων τις οποίες διαπραγματεύσαμε με μεγάλο μεγάλη δυσκολία τα τελευταία χρόνια και ελπίζω ότι συνεννοηθήκαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εφαρμόσει αυτά τα οποία συμφωνήθηκαν πέρυσι το Μάιο για το πακέτο τηλεπικοινωνιών. Βλέπω ότι ο Γενικός Διευθυντής ε, μιλά με τον Πρόεδρο, αλλά ελπίζω το μήνυμά μου να περάσει, δηλαδή ότι θα προσαρμόσετε και θα εφαρμόσετε αυτά τα οποία συμφωνήσαμε πέρυσι μετά από μακρές συζητήσεις, δηλαδή να υπάρξουν ε, ε, επενδύσεις εις τα δίκτυα νέας γενιάς μας εφόσον είχαμε σκεφτεί ε, πόσο τα δίκτυα αυτά της τρίτης γενιάς μπορούν να ενταθούν και τι χρειάζεται κατά τρόπον ώστε από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προχωρήσουμε ε, πέραν από αυτά τα οποία είχε προτείνει η Επιτροπή κατόπιν προτάσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ε, να μπορέσουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανταποκριθεί στις προσμονές ε, του Κοινοβουλίου διότι δεν θα θέλαμε η νέα Επιτροπή να παραβλέψει αυτά τα οποία είχαμε με προτείνει. Τώρα έχουμε μία νέα επιτροπή, μία νέα επίτροπο, αλλά ο Γενικός Διευθυντής ξέρει ακριβώς ότι ε, η συνθήκη της Λισαβόνας έχει εμπλουτίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ως εκ τούτου οι αποφάσεις του Κοινοβουλίου θα πρέπει επίσης να υλοποιούνται. Ευχαριστώ η κυρία Τικάου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα εδώ ε, να αναφερθώ σε αυτή την εξαιρετική έκθεση η οποία αποτελεί ένα σημείο εκκινήσεως όσον αφορά ε, την, ε, το σχετικό πρόγραμμα. Θα ήθελα όμως να κάνω μερικά σχόλια. Καταρχήν όσον αφορά την ε, οδηγία για τις υπηρεσίες, διότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να υπάρξει μία υπηρεσία από ένα κράτος μέλος θα πρέπει, δηλαδή δεν μπορεί ένα, μια τέτοια υπηρεσία να παράσχει υπηρεσίες σε ένα άλλο κράτος μέλος. Εφόσον λοιπόν μιλάμε για εσωτερική αγορά, θα έπρεπε να ανταποκριθούμε και σε αυτή την ανάγκη. Η ε, ψηφιακή λοιπόν αυτή ατζέντα ελπίζω ότι θα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων μας υλοποιήσεως και ολοκληρώσεως της ενιαίας αγοράς όσον αφορά τις αρμοδιότητες στα ψηφιακά θέματα και τις δεξιότητες. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να έχουμε μία κοινωνία της πληροφορικής εάν οι εμπλεκόμενοι δεν γνωρίζουν την τεχνολογία και οι χρήστες δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις τεχνολογίες. Πέραν αυτού χαιρετίζουμε το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές στο έγγραφο αυτό σχετικά με την πλήρη ευρυζωνική κάλυψη και αυτό αναφέρεται και στο πρόγραμμα οικονομικής ανακάμψεως, δηλαδή θα διατεθούν πόροι ε, για την ολοκλήρωση του προγράμματος αυτού μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Ως εκ τούτου η ε, προσφυγή ε, στα ψηφιακά συστήματα θα μπορέσει να ε, επιτρέψει ένα συνδυασμό των ε, τωρινών και μελλοντικών χρηστών οι οποίοι θα επωφεληθούν από αυτές τις εξελίξεις της ε, κοινωνίας της πληροφορικής. Όσον αφορά τώρα την ασφάλεια, θα ήθελα να σας πω ότι όντως όσον αφορά την, τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των ε, στοιχείων και της προσωπικής ζωής είναι βασικά θέματα αλλά πρέπει να υπάρχει και ε, εμπιστοσύνη των κατανολωτών ε, από πλευράς της κοινωνίας η οποία να βασίζεται στην εμπιστοσύνη που θα έχουν σε αυτές τις υπηρεσίες. Έχω προτείνει ορισμένες τροπολογίες και θα ήθελα να τονίσω πόσο σημαντική είναι η εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης διότι εδώ ε, θα πρέπει να μπορούν να γίνονται αγορές μέσω ηλεκτρονικών μέσων και τα Ηνωμένε Πολιτείε είχαν ε, υποσχεθεί ότι ε, το 2010 πέραν του 50% θα μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά αλλά απέχουμε πολύ από αυτό και ελπίζω ότι το πρόβλημα θα έχει επιληθεί μέχρι το 2015. Όσο αναφορά την ε, ε, την οδηγία για την τιμολόγηση η ε, νέα επίτροπος υποσχέθηκε να ασχοληθεί με το θέμα και κατόπιν μη ενός συνεδρίου την Άνοιξη ή στην Ισπανία να μπορέσει να επιτύχει την εφαρμογή των ηλεκτρονικών ε, τιμολογίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο διότι το κόστος για μία τέτοια διεκπαιρέωση θα μειωθεί κατά 10 ευρώ αναπερίπτωση, οπότε θα υπάρξει μία εξοικονόμηση πέραν των 500 εκατομμυρίων ευρώ. Άρα μεγάλο όφελος και για τον καταναλωτή αλλά και μείωση των δημοσίων εξόδων. Ε, όσον αφορά τις ε, αγορές του δημοσίου πρέπει να ε, λάβουμε υπόψη ότι είναι ένα μεγάλο μέρος του ΑΕΠ και είναι μια πολύ σημαντική αγορά άρα θα πρέπει να βοηθήσουμε εδώ τον ηλεκτρονικό αυτό τομέα διότι η, τα έξοδα αποτελούν το 11 μέχρι 18% των συνολικών συνολικών ε, ε, δημοσίων δαπανών. Δυστυχώς όμως αυτή τη στιγμή ε, στην Ευρώπη δεν υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφόρων δημοσίων υπηρεσιών, ιδίω αν πρέπει η υπηρεσία αυτή να παρασχεθεί ηλεκτρονικά. Η Γερμανία δεν μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες στη Γαλλία, διότι η νομοθεσία απαιτεί ένα πιστοποιητικό πολιτικό ψηφιακό που θα έχει εκδοθεί στη Γαλλία και αυτό είναι εφικτό μόνο για μέσω μιας εταιρείας η οποία να εδρεύει στη Γαλλία. Ευχαρίστως λοιπόν θα ήθελα να δω τα διάφορα προγράμματα που αναφέρονται στην αλληλεπίδραση των προγραμμάτων και στις αγορές ηλεκτρονικών μέσων ε, κάτι το οποίο ελπίζουμε ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2011 και από ό,τι ξέρω τον Οκτώβριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διατυπώσει ένα πρόγραμμα για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση προσβλέπουμε σε κάτι τέτοιο και θα ήθελα να πω ότι η ασφάλεια και η αλληλεπίδραση ε, όσον αφορά την ηλεκτρονική υπογραφή θα αποτελέσουν θέματα κλειδιά. Ε, τελειώνοντας παραπέμπω, ε, παραπέμπω στις έξυπνες πόλεις ή στους έξυπνους μετρητές για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε βελτιώσουμε την ποιότητα ζωή όλων των πολιτών της Ευρώπης. Συγχαίρω και πάλι την ηγήτρια και ελπίζω ότι η αυριανή ψηφοφορία πραγματικά θα δώσει ένα εναρκτήριο λάκτισμα σε προόδου στον τομέα της ψηφιακής ατζέντα. Ο κύριος Τσουκαλάς έχει τώρα το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα πήρα το λόγο για να ευχαριστήσω πρώτα την κυρία Πιλάρ καστίγιο Βέρα για την εξαιρετική της έκθεση καθώς επίσης και όλους τους συναδέλφους οι οποίοι με μεγάλη ε, προσοχή εξέτασαν ένα τόσο σημαντικό εργαλείο το οποίο το Ευρωκοινοβούλιο θέτει στη διάθεση ε, της Κομισιόν για την εφαρμογή πολιτικής. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι μιλάμε για το μέλλον της Ευρώπης, όπως αυτό θα διαμορφωθεί στην νέα κοινωνία, την κοινωνία του 21ου αιώνα, μεγάλο τμήμα των δραστηριοτήτων των πολιτών, καθώς επίσης και των δημοσίων οργάνων του, θα εξαρτάται από την τεχνολογία αυτή. Ήδη με την εξαγγελία της ε, Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών των Ηνωμένων Πολιτειών για το νέο σχέδιο σχετικά με την ευρυζωνικότητα και τις παροχές που ελπίζει η Αμερικανική Διοίκηση να δώσει στους Ευρωπαίους πολίτες καθώς και στα δημόσια σχολεία και τα ερευνητικά κέντρα τίθεται ήδη ο για την Ευρώπη ε, τον οποίον πρέπει να υπερπηδήσουμε εάν η πολιτική μας για το όραμα του 2020 είναι πραγματικά η αριστεία και εξακολουθεί να επιμένει ότι θα βασιστούμε στην κοινωνία της γνώσης. Σημείωσα ότι ε, οι συνάδελφοι ήταν ιδιαίτερως προσεκτικοί σχετικά με τους νέους και την ψηφιακή απομόνωση. Πράγματι, παρά τα αντιθέτως λεγόμενα, υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι η ψηφιακή απομόνωση αρχίζει και διαχωρίζει νέους από ηλικίε 17 χρονών, πράγμα που σημαίνει ότι τους κάνει λειτουργικά αναλφάβητους, πράγμα που είναι επίσης εξαιρετικά πιο ε, κακό παρά για κάποιον ο οποίος βρίσκεται στα σδισμά του επαγγελματικού του βίου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και ο τελευταίος ε, δεν πρέπει να βοηθηθεί. Το κακό είναι ότι δεν έχουμε μια πραγματική επανάσταση της ε, πληροφορικής. Επανάσταση νοείται όταν μια τεχνολογία τίθεται στη διάθεση του κάθε πολίτη άσχετα από τη μορφωτική του κατάσταση χωρίς την ιδιαίτερη γνώση οτιδήποτε άλλου. Για παράδειγμα, σήμερα οποιοδήποτε μπορεί να γυρίσει, να πατήσει ένα διακόπτη και να έχει ένα ηλεκτρικό ρεύμα. Μέχρι ότου η τεχνολογία της πληροφορίας βρεθεί σε αυτό το επίπεδο, θα χρειαζόμαστε να παίρνουμε μέτρα για να υποστηρίξουμε τους αδύνατους να καταλάβουν την τεχνολογία. Το πρωί ε, συζητήσαμε για ε, το ίντερνετ των πραγμάτων, δηλαδή για το FES περιβάλλον, το οποίο και είναι ίσως μια απάντηση με όλες τις επιφυλάξεις μας σχετικά με αυτά τα ζητήματα. Και πάλι να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για την προσοχή τους και ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρησιμοποιήσει αυτό το εργαλείο που ε, δίνει στη διάθεσή του το Ευρωκοινοβούλιο για την εφαρμογή αυτού του οράματος. Ευχαριστώ πολύ. Και τελευταίος ο κύριος Λάμπερτς. Λυπάμαι που άργησα λίγο. Ευχαριστώ που μου δώσατε το μικρόφωνο δεν θα το χρησιμοποιήσω για πολύ. Οι πράσινοι είχαν πει σε όλες τις προηγούμενες ε, συνεδριάσεις και στη σημερινή τα ίδια πράγματα. Ε, καταρχήν υπάρχει ανάγκη γρήγορης εργασίας. Πολλοί από εμά θέσαν ορισμένα θέματα επιτάπητος, οπότε φαντάζομαι ότι θα συμπεριλάβετε στον τρόπο εργασίας σας τα όσα είπαμε. Ε, θα, για την έκθεση τώρα την ίδια θέλω να αναφέρω τις ε, τροπολογίες ε, ε, στο, 90, 98 και συζητήσαμε για την τροπολογία 135, 138. νομίζω ότι πραγματικά δεν πρέπει να ξανανοίξουμε τη συζήτηση, δεν θέλω να το κάνω αυτό αλλά αυτή η παράγραφος, η παράγραφος 19 όπως επαναδιατυπώθηκε μιλάει αρκετά για την ανάγκη ισορροπίας για, για τη διάδοση της κουλτούρας μέσω του διαδικτύου και θα κρατούσα το 19 και το 19b ε, λέτε εκεί μιλάτε για την ε, λογική που διέπει την εξέβρεση ενός νέου μοντέλου ε, που να διέπει και τα πνευματικά δικαιώματα του συγγραφέα του και τα δικαιώματα του χρήστη. Αυτό είναι σωστό, δεν έχουμε τέτοιο πρότυπο. Είναι επίγον το καθήκον αυτό να εφεύρουμε ένα τέτοιο πρότυπο. Αλλά είναι αρκετά αυτά που λέγονται στο 19. Δεν χρειάζεται 19α ίσως να μπορεί κανείς να αναρωτηθεί περί τίνος πρόκειται, αλλά δεν χρειάζεται να ξανανοίξουμε τη συζήτηση πάνω σε αυτό το σημείο. Ε, για όλα τα υπόλοιπα ε, πρέπει να σας πω ότι συμφωνήσαμε και δεν θέλω να επαναλάβω τα όσα ήδη είπα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ θερμά και θα ήθελα να δώσω τέλος το λόγο εις ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Γενικό Διευθυντή Κολασάντη, αλλά ο κύριος Κολασάντη εδώ σε αυτήν τις θέσεις ε, έρχεται τελευταία φορά, διότι σε τρεις μέρες αποσύρεται και θα έχει ατελείωτο ελεύθερο χρόνο. Θέλω λοιπόν να τον ευχαριστήσω για την καλή συνεργασία που είχαμε κατά τους τελευταίους μήνες και τα τελευταία χρόνια όπου υπήρχαν συνεχείς ε, διενέξεις, διαμάξεις, ε, ε, διαμάχες αλλά και θετικά αποτελέσματα και γι' αυτό θα ήθελα να τον παρακαλέσω τώρα να μας βοηθήσει να οδηγήσουμε σε πέρα σε αυτό το πρόγραμμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για αυτά τα καλά σας λόγια. Ευχαριστώ για τη στήρεξη την οποία προσφέρατε σε μένα και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι πάντοτε τιμή για τους ε, υπαλλήλους Ευρωπαϊκής Ενώσεως να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί συμβάλλουν στην οικοδόμηση της Ευρώπης. Άρα θερμά ευχαριστήρια για τα καλά σας λόγια και την στήριξή σας θα εγκαταλείψω με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά θα παραμείνω σε ορισμένους τομείς που σας ενδιαφέρουν και μέχρι το τέλος του 2010 που ακόμη θα ε, εργάζομαι για την Ευρωπαϊκή Ένωση στα θέματα του διαδικτύου θα με ξανακούσετε. Αλλά ε, τώρα θα ολοκληρώσω και θα πω λίγα λόγια σχετικά με την έκθεση αυτή. Πρώτα απ' όλα ε, θα πω κάποια πράγματα για το χρονοδιάγραμμα, για τη διαδικασία και λίγα πράγματα για την έκθεση. Ε, τα πάντα οδεύουν όπως έχουν προγραμματιστεί. Η έκθεσή σας θα ψηφιστεί αύριο εδώ στην Επιτροπή και στη συνέχεια στην Ολομέλεια τον Απρίλιο, γεγονός που θα μας δώσει αρκετό χρόνο ώστε να λάβουμε υπόψη και τη συνεισφορά σα ε, στο έγγραφο το οποίο θα παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ψηφιακή ατζέντα και να διαβεβαιώσω την κυρία Νίμπλερ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει πάρα πολύ καλά πόσο σημαντικό γίνεται συνεχώς το Κοινοβούλιο και αυτό θα αντικατοπτρίζεται και στον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε, θα αναλύσουμε και θα λάβουμε υπόψη μα την ε, έκθεση που θα λάβουμε από το Κοινοβούλιο. Ε, να κάνω και δύο σχόλια για την έκθεση. Το ένα είναι για ένα σημείο το οποίο έχουν ήδη ανεφέρει αρκετοί από τους προλαλήσαντες, το που θα εστιάζει δηλαδή η έκθεση και το δεύτερο είναι αυτό το οποίο θεωρώ εγώ ίσως το πιο σημαντικό στοιχείο που έχει να προσφέρει η έκθεση αυτή το γεγονός δηλαδή ότι επισημαίνουμε τα αποτελέσματα, την κοινοτιμία και τη διακυβέρνηση ως προς το πού εστιάζει η έκθεση. Αυτό δεν ήταν ε, εύκολο σε καμία περίπτωση. Ε, το πλαίσιο, όπως πολύ σωστά το ανέφερε η κυρία Καστίγιο, ε, το οποίο καλύπτει η ψηφιακή ατζέντα, είναι πολύ ισχυρέ στις 18 Ιανουαρίου ε, εγκρίθηκε μία ανακοίνωση και παρουσιάστηκε από κοινού με την Ισπανική Προεδρία στη Μαδρίτη. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει και πάρα πολλές συστάσεις, γεγονός που καταδεικνύει πόσο σημαντικό είναι το θέμα αυτό και πόσο ευρύ είναι το πεδίο εφαρμογής που καλύπτει. Ε, εσείς έχετε καταφέρει να εστιάσετε σε κάποια σημεία στην ανάγκη να υπάρχει μια υποδομή, να υπάρχει μια ενιαία αγορά ως τρόπο ε, μέτρησης της πρόοδου που έχει επιτευχθεί και όπως είπατε και εσείς στην αρχική σας παρέμβαση, όλα αυτά με επίκεντρο το χρήστη, με τελικό στόχο το χρήστη ε, για όλα αυτά τα μέτρα που έχετε για τις δεξιότητες και ούτω καθεξής. Η έκθεση είναι πολύ πυκνή, περιλαμβάνει πολύ σημαντικά στοιχεία και μας δίνει και μία σειρά από χρήσιμα σημεία τα οποία θα ε, χρησιμοποιήσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να περάσω στη δεύτερη παρατήρηση μου όμως που θεωρώ ότι είναι και πιο σημαντική. Σαφώς ε, η κατάσταση όσον αφορά στην προαγωγή των ε, τεχνολογιών ε, πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, πόρα απέχει από αυτό που είχαμε πριν από 5 ή από 10 χρόνια. Η κατάσταση όλα είναι αλλαζει και οι τεχνολογίες συνεχώς εξελίσσονται. Αλλά η ανάγκη να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα, να έχουμε καλύτερες τεχνολογίες πληροφορίας και τηλεπικοινωνιών υπάρχει πάντα. Εδώ τώρα είναι και κατεπίγουσα η ανάγκη για την οποία χρειαζόμαστε αποτελέσματα. Και νομίζω ότι η έκθεσή σα επισημαίνει το γεγονό ότι ναι, έχουμε πει κάποια πράγματα επανειλημμένω, αλλά αυτή τη φορά ε, πρέπει να πούμε ότι τα χρειαζόμαστε και πρέπει να έχουμε αποτελέσματα. Χαιρετίζω και το θάρρος σας, διότι ζητάτε ε, πιο αποτελεσματικό benchmarking. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε κάποιο βαθμό έκανε και benchmarking στο παρελθόν, διότι πάντα χρησιμοποιούσαμε αναλύσεις, εκθέσεις για την απόδοση των κρατών μελών, αλλά σαφώς εσείς μας ενθαρρύνετε να προβληθεί αυτό πιο πολύ και να είμαστε και βέβαιοι ότι υπάρχει μια κάποια πίεση, η οποία είναι συλλογική και απευθύνεται προς όλους όσους έχουν την ευθύνη εφαρμογή των μέτρων. Και χαιρετίζω επίσης και το γεγονός ότι ε, εστιάσετε την προσοχή σας στην εφαρμογή όλης της νομοθεσίας μεν, αλλά κυρίως του ρυθμιστικού πλαισίου. Έχουμε πλέον κάποιους κανόνες, πρέπει να τους εφαρμόσουμε και υπάρχουν και πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι σε κρεμότητα. Ε, χαίρομαι λοιπόν για το γεγονός ότι ενδιαφέρεστε για αυτή την πτυχή. Είμαστε σε συζητήσεις και με την Ισπανική Προεδρία για να έχουμε ίσως στο επόμενο Συμβούλιο Τηλεπικοινωνιών μια συζήτηση επί του θέματος αυτό, επί τη βάση και δύο εκθέσεων που παρουσιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εφαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου και για την εφαρμογή ε, της διαδικασίας που γνωστή, ε, είναι γνωστή στην Ευρωπαϊκή Ορολογία ως τη διαδικασία του άρθρου 7. Σας ευχαριστώ λοιπόν, διότι και εσείς εστιάσατε στην εφαρμογή και στην επίτευξη των αποτελεσμάτων. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, έτσι ολοκληρώσαμε αυτή τη συζήτηση για σήμερα και την ε, ε, ολοκληρώσαμε για να μπορέσουμε αύριο να ψηφίσουμε. Ελπίζω δεν θα αλλάξουν άλλα πράγματα τη νύχτα. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον ε, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα έχουμε το επόμενο θέμα Internet New Governance Next Steps. Η κυρία Σούζα Βάγνερ είναι η μιλήτρια και της δίνω το λόγο για τη διακυβέρνηση του ίντερνετ τα επόμενα βήματα. Ο κύριος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επειδή η Επιτροπή μας είναι πολύ πλούσια και έχει και μία ποικιλομερφία θεμάτων, Ίσως θα πρέπει να σας υπενθυμίσω εδώ ε, το θέμα αυτής της έκθεσης. Η έκθεση αυτή αναφέρεται, όπως είπατε και εσείς, στη διακυβέρνηση του ίντερνετ και στην ανάλυση και στην κατάσταση ε, της κεντρικής φιγούρας που έχουμε παγκοσμίων για τη διακυβέρνηση του ε, ίντερνετ που είναι η ICAN. Η ICAN είναι μια οργάνωση sui generis, ε, μια μοναδική οργάνωση διότι διέπεται από αμερικανικό δίκαιο ή πιο συγκεκριμένα από το δίκαιο ε, μίας εκ των πολιτιών των ΗΠΑ γεγονός το οποίο δημιουργεί πάρα πολλές διαμαρτυρίες, πολλές επικρίσεις παγκοσμίω και είναι και πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι προτείνουν μία εκβάθρον αναθεώρηση αυτής της Αμερικανικής οργάνωσης. Υπάρχουν απόψεις ε, για όλα τα γούστα. Κάποιοι θεωρούν ότι αυτή η οργάνωση θα πρέπει να εξαφανιστεί, να μην ε, υφίσταται, επειδή ακριβώς είναι και μια ιδιωτική οργάνωση και να βρίσκεται μια νέα οργάνωση υπό την ε, σκέπη του ΟΗΕ. Και υπάρχουν και άλλοι ε, διεθνείς άλλες διεθνείς προτάσεις. Εμείς εδώ, το είδαμε και στην παρέμβασή μου την προηγούμενη φορά και στα όσα είπα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ξεκινάμε από αυτά που μας έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωσή της και θέλουμε να είμαστε υπέρ της διατήρησης αυτής της αμερικανικής οργάνωσης, αλλά ταυτόχρονα να προτείνουμε και μία εκβάθρον μεταρρύθμισή της. Εμείς ε, φρονούμε και εγώ αυτό θέλω να συμπεριλάβω στην έκθεση που προετοιμάζω ότι η ICAN χρειάζεται μεταρρύθμιση και χρειάζεται και πολύ σημαντικές ε, διορθώσεις. Ε, σας ευχαριστώ την προσοχή, συνάδελφοι. Εάν θέλουμε ο κυβερνοχώρος να είναι ένας χώρος ελευθερίας, νοτομίας και ευελιξίας, ένας χώρος το οποίο θα έχει την ικανότητα προσαρμογής, δεν μπορούμε ταυτόχρονα να θεωρούμε ότι η κεντρική οργανωτική δομή του, η ICAN δηλαδή, ε, να είναι μια ανελαστική και αμετακίνητη οργάνωση. Εάν ο κόσμος του ίντερνετ είναι δυναμικός, αυτός ο δυναμισμός πρέπει να εφαρμόζεται και στην ICAN. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, επιμένω, η ICAN είναι μια αμερικανική οργάνωση που αυτή τη στιγμή διαχειρίζεται τη διακυβέρνηση του ίντερνετ παγκοσμίω χρειάζεται μία πολύ έντονη απάντηση και αυτό ακριβώς θα προσπαθήσουμε να δώσουμε εμείς μέσω της έκθεσής μας ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εξ ε, του εισηγητή, θέλει να τονίσει ότι το ίντερνετ καταρχάς είναι ένα δημόσιο αγαθό. Ένα δημόσιο αγαθό του οποίου ο μονομορής έλεγχος από μία και μόνη κυβέρνηση δημιουργεί τεράστιες επικρίσεις, όπως σας είπα και πριν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει λοιπόν να αναπτύξει μία στρατηγική η οποία θα αντικατοπτρίζει ένα συνενετικό όραμα από όλε τις περιοχές του κόσμου για τις ε, βασικές πτυχές διακυβέρνησης του διαδικτύου. Τόσο τα διεθνή φόρα όσο και ε, στις ε, ε, διμερείς του επαφές με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να διαφαίνεται αυτό. Ο υποφαινόμενος θεωρεί ε, και με τα όσα λέει το, ε, η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι καλό θα ήταν ο ιδιωτικός τομέας να δραματίζει θεμελιώδη ρόλο στη διακυβέρνηση του διαδικτύου. Επειδή είναι τόσο μοναδικός ο τρόπος της διακυβέρνησης του διαδικτύου, έχουμε ιδιωτικά και δημόσια στοιχεία, έχουμε ιδιωτικά και ε, δημόσια υποκείμενα. Και εδώ ακριβώς είναι το νέο, το καινοτόμο στοιχείο της διακυβέρνησης του διαδικτύου. Με εφαλτήριο αυτό και ε, με τη σχέση με την ICAN προσπαθούμε, θα προσπαθήσουμε, αν εγκριθεί η έκθεση μάλλον, από την ICAN να συγκεκριμενοποιήσουμε τα νέα στοιχεία μεταρρύθμισης τα οποία έχουν δημιουργηθεί ε, στο ε, εσωτερικό της ICAN, διότι αυτά τα συγκεκριμένα μοντέλα θα μπορούν να αντιπροσωπεύουν τα, ε, διάφορα, τις διάφορες περιοχές του κόσμου, την ποικιλομερφία που έχει ο κόσμος και το πώς ενδιαφέρεται με το, για το διαδίκτυο ο κόσμος. Στόχος μας λοιπόν θα είναι να δοθούν κίνητρα ώστε να ενεργοποιηθούν όλοι οι μηχανισμοί που θα βρίσκονται στα νέα μέτρα αναθεώρησης που θέλει να ε, κάνει η δομή της ICAN. Δεύτερον, θα ήθελα να τονίσω πόση σημασία έχει το ε, GAC που είναι η Συμβουλευτική Επιτροπή των Κυβερνήσεων της ICAN ε, πρόκειται για ένα συμβουλευτικό όργανο το οποίο εκδίδει συστάσεις και θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος του ώστε να επιτρέπεται μέσω αυτής της οδού να συμμετέχουν στη διαχείριση του διαδικτύου οι διάφορες γεωγραφικές περιοχές στις οποίες απευθύνεται ο κυβερνοχώρος και το διαδίκτυο. Επίσης, θα πρέπει να διατηρήσουμε και την εθνική ταυτότητα των ε, ε, μελών, των υπαλλήλων, του προσωπικού που είναι στην ε, υπηρεσία της ICAN. Θα πρέπει να αναλύσουμε και τους πόρους από τους οποίους χρηματοδοτείται το ICAN αυτή τη στιγμή. Η, αυτή τη στιγμή οι πόροι είναι κυρίως αμερικανικοί Επομένω, επομένως η χρηματοδότηση θα πρέπει ίσω να ανοίξει για να διαφοροποιηθεί και να μην έχουμε ανεπιθύμητες κυρίαρχες θέσεις λόγω του τρόπου χρηματοδότησης. Ξεκινώντας λοιπόν από την οργάνωση αυτής τη οργάνωση που επαναλαμβάνω ότι είναι αμερικανική, θεωρούμε ότι θα πρέπει να παραμείνει το φόρουμ συζήτησης του διαδικτύου, που είναι το φόρουμ διακυβέρνησης του διαδικτύου. Αυτό το φόρουμ λοιπόν για τη διακυβέρνηση του ε, διαδικτύου αποδείχθηκε μεγάλη επιτυχία, διότι εδώ ε, έχουμε συγκερασμό απόψεων από όλους τους ενδιαφερομένους και μάλιστα με ελεύθερο και παραγωγικό και γόνιμο τρόπο, όταν βλέπουμε και τις ε, πράξεις που προκύπτουν από όλα αυτά, ε, ασχολήθηκε με όλα τα θέματα τα οποία αφορούν αυτόν τον κόσμο ο οποίος είναι τόσο σημαντικός. Υπάρχουν βέβαια μια σειρά από διορθώσεις που θα πρέπει να γίνουν στη λειτουργία αυτής της οργάνωσης, αυτού του φόρουμ και εγώ ε, προσπάθησα να τα επισημάνω εδώ σε αυτό το έγγραφο εργασίας. Σας έχει διανεμηθεί άλλωστε το έγγραφο εργασίας και εδώ θεωρούμε και αυτό προτείνω κιόλας ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ε, ε, θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ισπανικής και Βελγικής Προεδρίας στο Βίλνιους όταν θα συγκληθεί η επόμενη σύνοδος κορυφής αυτού του Διεθνούς ε, Φόρουμ. Οι συνάδελφοι που με ακούν γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι το διαδίκτυο είναι ένας χώρος όπου καθημερινά υπάρχουν ειδήσει. Ε, καθημερινά όλες οι εφημερίδες ανά τον κόσμο συλλέγουν πάρα πολλές πληροφορίες που αφορούν αυτό το συγκεκριμένο χώρο, το διαδίκτυο. Υπάρχουν λοιπόν μια σειρά από θέματα τα οποία έχουν προκύψει από αυτή την έκθεση αλλά έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και είναι ε, προφανές ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά έργανα θα πρέπει να ασχοληθούν με τα θέματα αυτά. Ε, το κάνουν ήδη. Ακούσαμε σήμερα εν μέρη και το έγγραφο το οποίο εκπώνησε η κυρία Καστίγιο, αλλά υπάρχουν και άλλα έγγραφα εντός των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων που ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Όπως για παράδειγμα το να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει πρόσβαση για όλους χωρίς καμία διάκριση στο διαδίκτυο, κάποια στοιχεία που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια για απειλές ή επιθέσεις, την προστασία της ιδιωτικής ζωής, την ε, προστασία των ε, πνευματικών δικαιωμάτων και την ε, πρόσβαση για όλους τους χρήστες, να, την καταπολέμηση του εγκλήματος και την προάσπιση των δικαιωμάτων των ανηλίκων. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία όπως σας είπα είναι συνεχώς στις εφημερίδες, στον τύπο και συνεχώς κυκλοφορούν σε πάρα πολλά έγγραφα στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Σε αυτή την περίπτωση, ε, στην έκθεση που προσπαθώ εγώ να ετοιμάσω, τα θέματα αυτά ε, αναφέρονται με παρεπομπές ε, σε όλα τα υπόλοιπα έγγραφα τα οποία έχουν εγγραφεί, εγκριθεί είναι σε φάση έγκρισης, διότι ο δικός μας ο ρόλος είναι να ε, δούμε το πρόβλημα της διακυβέρνησης του διαδικτύου ε, και των οργανωτικών δομών που είναι στην υπηρεσία αυτής της διακυβέρνησης. Επιτρέψτε μου εδώ να τονίσω ότι ε, κατά την άποψή μου Καλό θα ήταν να υποστηρίξουμε την πρωτοβουλία της Ισπανικής Προεδρίας, να ετοιμάσει λοιπόν μια ευρωπαϊκή χάρτα των δικαιωμάτων των χρηστών του διαδικτύου καθώς επίσης και την ε, πρόταση να αναγνωρίσουμε την πέμπτη θεμελιώδη ελευθερία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που είναι η πρόσβαση στο διαδίκτυο. Όσον αφορά στην οργάνωση και την εσωτερική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να προχωρήσουμε θέματα που αφορούν στο συντονισμό μεταξύ των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων και την ICAN, η οποία δεν γίνεται πάντα με τον πιο λογικό τρόπο. Οι σχέσεις ε, ε, της Ευρώπης, των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων με αυτό τον αμερικανικό οργανισμό, την ICAN, δεν είναι πάντα οι κλασικές σχέσεις ε, διοικητικής λογικής. Γιατί? Γιατί κάποιες φορές υπάρχει έλλειψη συντονισμού μεταξύ της δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Συμβουλίου ή και του ίδιου του Κοινοβουλίου και της ICAN. Ε, καλό θα ήταν λοιπόν να προσπαθήσουμε να συνενώσουμε τις τάσεις μας και να δίνουμε ε, το συντονισμό των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων όσον αφορά τις σχέσεις της με την ICAN. Και τέλος θα ήθελα να επιμείνω στο γεγονός ότι η διακυβέρνηση του διαδικτύου, το θέμα δηλαδή που απασχολεί την έκθεση που σας παρουσιάζω, είναι μια πάρα πολύ σημαντική ευκαιρία ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να είναι παρόν και να προασπίσει το ε, προσωπικό του όραμα για τη διακυβέρνηση του διαδικτύου και τις αξίες του για αυτό το τόσο σημαντικό κεφάλαιο με μία φωνή στο διεθνές προσκήνιο. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο μπορεί να αποτελέσει προβολή της Ευρώπης και θα μπορέσουμε ίσως να δούμε την Ευρώπη να ε, μιλά με μία φωνή στα διεθνή φόρουμ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Τικάου έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε εν ονόματι της ε, Κατρίν ε, Τροτμάν που είναι η σκιώδης εισηγήτρια της πολιτικής μας ομάδας και δεν παρίσταται σήμερα θα παρουσιάσω την άποψή της. Θα ήθελα να ευχαριστήσει τον ε, εισηγητή, τον κύριο Σώσα Βάγνερ για το έγγραφό του που μπορεί να βοηθήσει ε, και αυτούς από εμά και εκτός του Κοινοβουλίου να κατανοήσουν σωστά την κατάσταση και να ε, γνωρίζουν ποιες είναι οι επιλογές τις οποίες έχουν. Υπάρχουν ε, ορισμένα ασαφή σημεία επί των οποίων θα προτανθεί στο κύριο Βάγνερ ε, με ηλεκτρονικό μήνυμα κατευθείαν θα ήθελε να στηρίξει την μέχρι τώρα προσέγγιση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων να βελτιώσουν ε, ε, την ισχύουσα οργάνωση της ICAN και εξηγεί γιατί οι άλλες εναλλακτικές λύσεις δεν είναι αποδεκτές διότι ε, ούτε το διακυβερνητικό σύστημα ούτε η πλήρης ε, ε, ιδιωτικοποίηση θα ικανοποιήσουν διότι πρέπει να συντονίσει κανείς τους πόρους και ουσιαστικά να εξετάσει επί καθημερινής βάσεως τα θέματα προς την διεθνή κοινότητα και προς το δημόσιο συμφέρον και τους καταναλωτές διεθνώς. Καλό θα ήταν εάν μπορούσαμε να επιτύχουμε ε, να βρούμε κάποιο τρόπο να συζητήσουμε την λειτουργία ΙΑΝΑ. Η κυρία Τροτμάν επιπλέον θα ήθελε να πει ότι ναι μεν βασιζόμαστε στην ΆΙΚΑΝ αλλά δεν είναι η μονατική δομή. Υπάρχουν και άλλες δομές οι οποίες ε, είναι πιο ικανοποιητικές όπως ε, η IATF και η ICOC. Τέλος, η κυρία Τράουτμαν θεωρεί ότι υπάρχουν ε, τρόποι να βελτιώσει κανείς τις ε, πλατφόρμες ε, μέσω ε, μιας ε, ευρωπαϊκής συνελεύσεως και ελπίζει ότι το έγγραφο αυτό θα μπορέσει να αιτιολογήσει μια υξημένη εμπλοκή όλων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων για να βελτιωθούν για να βελτιωθεί η πρόθεση στα διάφορα διεθνή όργανα ε, έχοντας μία σαφή προσέγγιση διότι διαφορετικά όλες οι αποφάσεις θα λαμβάνονται ρήμην μας. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω κανένα να ζητά το λόγο, οπότε θα ήθελα να δώσω τον λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριμένα στον κύριο Νίμπλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την έκθεσή του. Συμφωνούμε πλήρως ότι είναι ένα πολύ βασικό θέμα που αναφέρεται σε πολλούς τομείς του δικαίου. Μιλάμε για διανοητική ιδιοκτησία, για προστασία δεδομένων και όλα τα θέματα που θίξαμε και συμφωνούμε ότι πρόκειται για ένα global public resource και δεν μπορεί το θέμα αυτό να επιληθεί με ε, τον τρόπο που προτείνει η κυρία Τροτμάν μέσω της λειτουργίας ΙΑΝΑ. Εμείς συμφωνούμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε και ότι οι κυβερνήσεις μέσα στην ΆΙΚΑΝ έχουν μόνο μία συμβουλευτική μορφή. Το Α είναι κεφαλαίο, το advisory. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια δυνατότητα να προχωρήσει κανείς και αυτό τονίζεται στη γνωμοδότηση. Τέλος αυτό το φόρουμ για την διακυβέρνηση του ίντερνετ είναι πολύ σημαντικό διότι βλέπουμε ότι ε, ε, εκδηλώνεται σε ε, διάφορες εκδηλώσεις βελτίωση και την εικόνα που προβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά από τον πρώτο γύρο το φόρουμ αυτό ο πρώτος γύρος ολοκληρώνεται τώρα θα αποτελέσει μία νέα μορφή και τέλος όσον αφορά την accountability συμφωνώ με τον κύριο Σάντι ότι πρέπει να προχωρήσει. Ο εισηγητής ε, ε, Σόσα Βάγνερ ε, βασίζεται εις την επιβεβαίωση των δεσμεύσεων όπως είπε και αυτό αναφέρεται εις την συμπεριφορά των εμπλεκομένων. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μία βελτίωση σε τέσσερις τομείς. Ε, καταρχήν στην ε, διαφάνεια και ε, την απόδοση λογαριασμών όπως ανέφερε ο κύριος Σόσα Βάγνερ. Πρόκειται για μια βασική εξέλιξη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τη γίνηση αυτή. Θα ήθελα όμως να σας πω ότι ατυχώς δεν μπορώ να πω ότι οι ομάδες αναθεώρησης που έχουμε καταρτήσει για να παρακολουθούν την έκθεση αυτή σαν, ε, μπορούν να λειτουργήσουν σαν μηχανισμός ελέγχου όπως λέτε στην έκθεση αλλά ελπίζουμε ότι θα περάσουν θετικά τη διαδικασία διότι θα μπορέσουν να διατυπώσουν ε, συστάσεις και ούτω καθεξής. Ζητήσατε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι ενεργή, να ε, μπορέσει να διασφαλίσει την ανεξαρτησία των διαφόρων μελών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υπάρξει ενεργή ε, και όπως είπα συζητήσαμε και με τα κράτη-μέλη έχουν ε, ε, στα πλαίσια τύπων ε, συνεδριάσεων και προς το τέλος του παρελθόντος έτους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε ένα πρώτο βήμα, πρότεινε έναν εθελοντή για μία από αυτές τις ομάδες όσον αφορά την ε, ε, διαφάνεια και την ε, απόδοση προσεφέρθη η κυρία Ρέντινγκ να συμμετέχει σε αυτή την ομάδα και χθες δημοσιεύτηκαν οι αιτήσει τις οποίες είχαμε ζητήσει και ελπίζουμε ότι θα έχουμε σύντομα τη σύσταση και τον Απρίλιο θα θα μπορέσουν να αρχίσουν οι εργασίες με όλους τους ενδιαφερόμενους και θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του χρόνου. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σούζα Βάγνερ νομίζω ήθελε ακόμη να πει δύο πράγματα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να πω απλώς ότι ευχαριστώ πολύ για τα τόσο καλά λόγια που άκουσα για τη δουλειά μου. Να πω ότι οι παρατηρήσεις που μου κάνει η κυρία Τράουτμαν θα ληφθούν υπόψη ε, σίγουρα ε, διότι άλλωστε γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα θέματα αυτά ε, και έχει ασχοληθεί με αυτά εδώ και πάρα πολύ καιρό και ε, εκτιμώ και ιδιαίτερως όλα όσα ακούσαμε από τις εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα και το να ασχολείται κάποιος με ένα θέμα όπως είναι αυτό είναι εξαιρετικό διότι καθημερινά υπάρχουν νέες ειδήσει, νέα στοιχεία και θα πρέπει να είμαστε σε γρήγορση να παρακολουθούμε τον τύπο και να βλέπουμε τι ακριβώς λέει. Είναι πιθανό όταν ψηφιστεί το, η έκθεση, όπως ε, προβλέπετε, να έχουν προκύψει και μια σειρά από γεγονότα τα οποία θα πρέπει να μας ε, ε, κάνουν να αλλάξουμε τη θέση μας. Αλλά αυτό είναι συνέπεια του να ασχολούμαστε με ζωντανά θέματα, διότι το θέμα αυτό είναι καθόλου ζωντανό, δεν έχει πεθάνει σε καμία περίπτωση. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να εργαστούμε και να συνεχίσουμε να εκπονούμε αυτό το ψήφισμα. Να πω επίσης ότι η δική μου η δουλειά δεν θα μπορέσει να είναι παρά ένα λιθαράκι, ε, διότι πολύ μεγάλη δουλειά έχει γίνει και από τους ε, συνεισηγητές, τους κοιόδης συγητές που εργάστηκαν για το θέμα αυτό και ελπίζω να κάνουν το ίδιο και για το πρόταση ψηφίσματος να σας ανακοινώσω εκ των προτέρων, αν και νομίζω ότι αυτό υπάρχει και στα έγγραφα που σας ε, ε βγαίνει με η γραμματεία, στις 4 Μαΐου θα κάνουμε μία ακρόαση με τους εμπειρογνώμονες που έχουν προταθεί, οι περισσότεροι από τους συνεισηγητές και μπορούμε ε, να συζητήσουμε μαζί τους και να ανταλλάξουμε απόψεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συμπληρώσω ότι 6 Μαΐου είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες. Και τώρα ερχόμαστε στο επόμενο θέμα, αριθμός 9, διασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην εσωτερική αγορά. Η συγητής είναι ο κύριος Πάουλ Ρούμπιχ και έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε ε, Πρόεδρε Ρόιλ η διανοητική ιδιοκτησία και το copyright είναι θέματα τα οποία μας απασχολούν πάρα πολύ διότι οι διεθνείς ταχύτητα των επικοινωνιών έχει αυξηθεί πάρα πολύ και εδώ δεν αναφερόμαστε μόνο στις τεχνικές δυνατότητες μεταφοράς περιεχομένου που γίνονται όλο και πιο σημαντικές αλλά και την μετάδοση στοιχείων μέσω του διαδικτύου και των τεχνικών δυνατοτήτων οι οποίες υπάρχουν. Δεν αναφερόμαστε μόνο στις τεχνικές βάσεις αλλά και στο περιεχόμενο και ποιο περιεχόμενο ε, κατόπιν αυτού μπορούν ε, να ε, ρυθμιστούν και να προσφερθούν σωστά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ε, με μία ε, ουδέτερη αντιμετώπιση τεχνολογική κατά τρόπον ώστε όλοι να μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες υπό τους ίδιους όρους. Γι' αυτό χρειάζεται ε, μία συλλογική διακήρυξη των δικαιωμάτων στην Ευρώπη και γι' αυτό αποφασίσαμε να εισάγουμε την ιδέα του One Stop Shop, δηλαδή για αυτόν ο οποίος θέλει να δημιουργήσει το περιεχόμενο και αυτό που θέλει να το χρησιμοποιήσει να είναι πιο απλό και πιο διάφανο το σύστημα το οποίο ισοσκελημένα να μπορεί να υποστηρίξει την προσπάθεια. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορέσει να βρεθεί μία ρυθμισμένη λύση. Εξού και από την European Broadcasting Union εχθές και σήμερα είχαμε μία πολύ σημαντική παρουσίαση διότι θέλουμε να δώσουμε νέες δυνατότητες και πρέπει να απευθύσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το σύστημα αυτό να διαμορφωθεί με διαφάνεια και απλά. Όσον αφορά τη διανοητική περιουσία ε, βρισκόμαστε σε μια εσωτερική αγορά. Δεν πρέπει να υπάρξουν φοβερές ε, γραφειοκρατικές δυσκολίες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα πρέπει για τους καταναλωτές, για τους πολίτες να δοθεί η δυνατότητα να χρησιμοποιούν τη δικιά τους γλώσσα σε όλες τις υπόλοιπες ε, χώρες της Ευρώπης χωρίς να υπάρχουν περίπλοκες απαγορεύσεις και νομοθεσίες που δεν επιτρέπουν στον Ευρωπαίο πολίτη σε μία ξένη χώρα να μπορεί να λάβει τα αναγκαία στοιχεία στην ε, γλώσσα του. Νομίζω ότι αυτό είναι μία βασική αρχή των γλωσσών μας. Έχουμε 23 γλώσσες, κάθε μία έχει τις ιδιομορφίες της και εγώ θα ήθελα απλώς σαν Γερμανός όταν βρίσκομαι στην Ισπανία παραδείγματο χάρη να μπορέσω να ακούω μια γαλλική εκπομπή και αν είμαι στην Ουγγαρία θα ήθελα να μπορώ να δέχομαι μία Ιταλική εκπομπή και νομίζω ότι ο πολίτης ε, έχει δικαίωμα να απαιτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, ε, λαμβάνει και να καταναλώνει το περιεχόμενο το οποίο παράγεται στη γλώσσα του σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε από πλευράς πολιτιστικής ταυτότητος πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι ο καθένας θα μπορέσει να έχει το διανοητικό περιεχόμενο είτε πρόκειται για εκπομπή η οποία είναι γραμμική ή όχι ε, θα πρέπει ο κάθε πολίτης να μπορεί να λάβει όλο το περιεχόμενο στη γλώσσα του σε ολόγινο κλήρη την Ευρώπη χωρίς να καθίσταται παράνομος. Νομίζω ότι βρήκαμε πολύ καλές λύσεις εδώ και εγώ είμαι διαθέσιμος στη συζήτηση να σημειώσω αλλαγές και αύριο να υποβάλω κατά την ψηφοφορία προφορικές τροπολογίες διότι πρέπει να παρουσιάσουμε μία γνωμοδότηση η οποία θα αποτελέσει τον πύχη με τον οποίο θα κριθεί η περαιτέρω εξέλιξη της Ευρώπης και οι συζητήσεις που είχαμε μεταξύ μας ήταν επικοδομητικές. Θέλω να ευχαριστήσω όλες τις πολιτικές ομάδες για την επικοδομητική συζήτηση και ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε μια θετική λύση. Ευχαριστώ. Έχει κάποιος κάποια δήλωση, η κυρία Τικάου. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα ε, ο ως να ε, ευχαριστήσω τον κύριο Ρούμπικ, συντάκτη της ε, εισήγησης, ειδικά για τα όσα είπε μέσα σε αυτήν την έκθεση που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, είναι αμέσω επίκαιρο ενδιαφέροντος. Θα ήθελα λοιπόν να υπογραμμίσω το γεγονός ότι οι άδειε σε ευρωπαϊκό επίπεδο που προσφέρουν ευρωπαϊκή κάλυψη μπορούν να συζητηθούν μόνον εφόσον θα έχουμε μια στήριξη για τις επιπτώσεις γιατί θα πρέπει να πάρει μέρος ο, ε, κάθε φορά ο αντίστοιχος βιομηχανικός τομέας. Ε, το ίδιο πράγμα ίσχυσε και για τον κινηματογράφο και για τη μουσική και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και για παράδειγμα. Θα πρέπει επίσης να επιστήσω την προσοχή σας στην παράγραφο 2 όπου γίνεται λόγος ε, για τις άδειες που βασίζονται στις ε, γλώσσες. Γίνεται η διάκριση με κριτήριο τη γλώσσα. Εδώ υπάρχει τροπολογία αριθμός 6. Αυτή η τροπολογία προτείνει να δοθεί ενδεχομένως η δυνατότητα να γίνονται υπότιτλοι για να μπορεί να υπάρχει σε περισσότερες ή ντουμπλάρισμα για να υπάρχει εκδοχή σε περισσότερες από μία γλώσσες. Ο κύριος Ρούμπικος θα μπορούσε να δεχτεί μια προφορική τροπολογία πάνω σε αυτό και στην αρχική τροπολογία αριθμός 6 θα ήθελα να προσθέσω κάτι ως, για όλους τους καταναλωτές δίνοντάς τους ε, ε, πρόσβαση στην γλώσσα παραγωγής και κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αντικατοπτρίσουμε και τα, το ενδιαφέρον των καταναλωτών που μπορεί να θέλουν να έχουν πρόσβαση στην ε, γλώσσα προέλευσης αλλά να υπάρχει το ε, ενδεχόμενο άλλων γλωσσών χωρίς να υπάρξει καινούρια άδεια που να βασίζεται στη γλώσσα όπου το κριτήριο να είναι μόνο γλωσσικό και αυτό ε, είναι πολύ σημαντικό σε σχέση με τους νόμους που διέπουν το μονοπόλιο. Οι μικρότερες γλώσσες ε, ε, μπορεί να έχουν πρόβλημα σε επίπεδο διανομής. Η αγορά των αδειών θα πρέπει να γίνεται γενικά χωρίς ανάγκη προσαρμογής των μικροτέρων γλωσσών και δεν υπάρχει και ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα των γλωσσών μίζωνων και λασών. Η κάθε χώρα έχει τη δική της πολιτική. Έχουμε όλοι γλώσσες εργασίας, γλώσσες μειονοτικές, αλλά στην περίπτωση αυτή το θέμα γίνεται πολύ λεπτό. Και γι' αυτό θα ήθελα να προτείνω και μια άλλη τροπολογία. Με την έγκρισή σας θα ήθελα να καταθέσω μια προφορική τροπολογία στην αρχική. Συγκεκριμένα, για τα θέματα των πνευματικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφόρησης δυστυχώς και επειδή έχουμε ορισμένες εξαιρέσεις οι οποίες αρμηνεύονται διαφορετικά από τα κράτη-μέλη φτάνουμε σε ένα σημείο όπου σε ορισμένες χώρες έχουμε ένα νόμο που ασχολείται με διαφορετικό τρόπο για ίδια φαινόμενα. Ε, δεν είναι μόνο διαφορές μεταξύ χωρών. Οι εταιρείε είναι πολυεθνικές ε, πάρα πολύ συχνά. Χρειάζεται λοιπόν μια ισχυρή νομική βάση και μια νομική βεβαιότητα. Χρειάζεται να γίνει λοιπόν μια αναθεώρηση της οδηγίας που αφορά τα πνευματικά δικαιώματα στην κοινωνία της πληροφόρησης για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Θα υποβάλω μια προφορική τροπολογία σχετικά και ε, θα χρησιμοποιήσω την διατύπωση πάνω στην οποία συμφωνήσαμε και ψηφίσαμε μάλιστα και επ' αυτής ε, πριν να ψηφίσουμε για την νέα Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είχε γίνει μια συζήτηση μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τότε, εάν θυμάστε. Λοιπόν, πέρα από αυτό, ε, νομίζω ότι ο εισηγητής ε, σίγουρα μπόρεσε να καταρτήσει ορισμένες συμβιβαστικέ τροπολογίες ε, που προστατεύουν τα δικαιώματα του χρήστη και ταυτόχρονα δεν μας επαναφέρουν σε πρώτερα κεφάλαια, δηλαδή κεφάλαια όπως είναι αυτά που αφορούν ε, τους κανονισμούς ε, που ισχύουν στον τομέα, στο πεδίο των ε, Telecom. Εν πάση περιπτώσει τα δικαιώματα του χρήστη πρέπει να προστατευθούν στην κοινωνία της πληροφόρησης. Η ασφάλεια του καταναλωτή, η πρόσβαση στα ιδιωτικά δεδομένα και η προστασία του ιδιωτικού βίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, η Κάριν. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο για όση δουλειά έκανε για το θέμα αυτό. Είναι ένα πολύ ακαθόδε ζήτημα το να προσπαθεί δηλαδή κάποιος ε, να βρει μια κάποια νομοθετική πρόταση για αυτό το θέμα και νομίζω ότι αυτή θα είναι μία από τις μεγάλες προσκλήσεις που θα αντιμετωπίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη διάρκεια της αιτίας αυτής. Ε, πολλοί συναδελφοί το συζητούν σε πολλές επιτροπές και είναι πολύ δύσκολο να βρούμε ένα νομοθετικό πλαίσιο για έναν τομέα ο οποίος εξελίσσεται με αλματώδη βήματα και ε, συνεχώς ε, μετακινείται ο πύχης. Εμείς λοιπόν ως Κοινοβούλιο θεωρώ ότι πρέπει να προχωρήσουμε το θέμα αυτό όσο το δυνατόν πιο ευρύτερα και να προσπαθήσουμε να προσφέρουμε ένα νομικό πλαίσιο το οποίο δεν θα είναι παρεχημένο ήδη από την ημέρα που θα οριστικοποιηθεί. Το νομικό πλαίσιο θα πρέπει να είναι ένα πλαίσιο το οποίο θα μπορεί να εξελίσσεται με τις ε, εναλλασσόμενες καταστάσεις, στο μέτρο του δυνατού φυσικά και καταλαβαίνω πόση δυσκολία υπάρχει για τον εισηγητή για να μπορέσει να έχει ένα ε, πλαίσιο το οποίο θα είναι ε, αποτελεσματικό από αυτή την έννοια. Να συγχαρώ λοιπόν τον κύριο Ρούμπικ και συμφωνώ ότι έχει αναλάβει ε, και μας έχει παρουσιάσει κάποια εξαιρετικά στοιχεία. Υπάρχουν δύο-τρία πράγματα τα οποία θα ήθελα να θίξω παρόλα αυτά ε, κυρίως ως προς τις ε, τροπολογίες που έχουν ε, κατατεθεί και θα ψηφίσουμε. Οι τροπολογίες 5, 6 και 2 κάνουν μία διάκριση μεταξύ εμπορικών παραποιημένων προϊόντων και μη εμπορικών παραποιημένων προϊόντων. Νομίζω ότι αυτό είναι μία τεχνική διάκριση, τουλάχιστον για μένα. Και μάλλον περιπλέκει τα πράγματα και δεν ε, προσθέτει κάποιο νέο στοιχείο στα όσα πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα της παραποίησης, της πειρατείας, με τον οποιονδήποτε τρόπο εκδηλώνεται. Ε, σαφώς ε, θα πρέπει να υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, αλλά το να κάνουμε μια τέτοια διάκριση δεν νομίζω ότι ε, μας ε, οδηγεί προς τη σωστή κατεύθυνση. Η τροπολογία 25 τώρα. Δέχομαι ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να, ε, σταματήσουμε, να προσπαθήσουμε να κινούμαστε προς ένα εναρμονισμένο σύστημα, πιο εναρμονισμένο αρχικός και τελικά πλήρως εναρμονισμένος. Αλλά σας εφιστώ την προσοχή εδώ, δεν θα πρέπει να ε, περάσουμε απευθείας στην ε, πλήρη εναρμόνιση. Και εδώ θα συμφωνήσω με τα όσα είπε και η συνάδελφός μόλις πριν από μένα, θα πρέπει να γίνεται αξιολόγηση και να υπάρχουν και αξιολογήσει αντικτύπου, διότι μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να δούμε πού ακριβώς βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και τι ενδέχεται να συμβεί σε θέματα τεχνολογικής προόδου τις επόμενες εβδομάδες, μήνες ή και χρόνια. Διότι η ταχύτητα με την οποία κινείται η τεχνολογία για να βοηθήσει τους ανθρώπους να διεξάγουν τη ζωή τους είναι εκπληκτική. Είναι λοιπόν θεμελιώδη σημασία να γίνει κάτι τέτοιο. Και τέλο έχουμε και μια τροπολογία την οποία κατέθεσα εγώ, την τροπολογία υπαριθμών 15, στην οποία ζητώ αποτελεσματικέ δράσει και όχι αποτελεσματικέ κυρώσει. Και δεν το ζητώ αυτό γιατί έχω κάτι εναντίον των κυρώσεων αυτών καθεαυτών. Το σκεπτικό μου είναι ότι χρησιμοποιώντας τον όρο δράση, όχι μόνο επιτρέπουμε να υπάρχουν και κυρώσεις, αλλά είμαστε και υπέρ της ε, ενεργούς δράσεις. Ε, δημιουργούμε το κατάλληλο περιβάλλον ώστε να μπορέσει να προχωρήσει και η βιομηχανία. Να σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα. Ε, προσφάτως συναντήθηκα με τον αρμόδιο φορέα ε, σε θέματα πνευματικών δικαιωμάτων ε, και παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών για τους κρυφείς στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και μου είπανε ότι σχεδόν όλες οι εμπορικές συναλλαγές παραποίησης γίνονται μέσω πιστοτικών καρτών λίγα πράγματα μπορούμε να κάνουμε με δράσεις για να μπορέσουμε να ε, σταματήσουμε αυτές τις χρήσεις και να απαγορεύσουμε σε κάποιον να κάνουν αυτές τις τόσο λανθασμένες και σε ορισμένες περιπτώσεις εγκληματικές πράξεις. Οι κυρώσεις από μόνες τους δεν αρκούν πρέπει να μπορούμε να κάνουμε και κάτι επιπλέον. Ε, να κρατήσουμε και την πτυχή των κυρώσεων, αλλά να υπάρχουν και κάποιες δράσεις επιπλέον. Ε, υπάρχουν πράγματα, υπάρχει περιθώριο να γίνουν περισσότερα πράγματα, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο το οποίο θα ενθαρρύνει τον ίδιο τον τομέα να κάνει ο ίδιος περισσότερα πράγματα για να βοηθήσει τον εαυτό του, αλλά και να βοηθήσουμε αλλήλους, να συνεργαστούμε και να επισημάνω για άλλη μια φορά ότι χρειαζόμαστε περαιτέρω αξιολόγηση και ε, αποτιμήσεις αντικτύπου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Έντσο έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να χαιρετήσω την έκθεση του κύριου Ρουμπίκ και την πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ενισχύσει την εφαρμογή των δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πραγματικά αυτό το θέμα και προκαλεί πολλές συζητήσει. Η συζήτηση δεν έχει ακόμα τελειώσει και μπορεί να συνεχιστεί και μετά από την έγκριση της παρούσας έκθεσης. Θα ήθελα να τονίσω μία μόνο πλευρά, ε, ένα θέμα με απασχολεί, ε, τους, ε, το ότι ε, όσοι παρέχουν ίντερνετ δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να είναι υπεύθυνοι για τις πράξεις των πελατών τους και θα πρέπει να μην είναι ε, υποχρεωμένοι να ασκούν επιθεώρηση. Δηλαδή επιθεώρηση παραδείγματο χάρη για λαθρεμπόριο που γίνεται μέσω του διαδικτύου κτλ. Ε, ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί σύνδεσμοι που ασχολούνται με τέτοια θέματα και υποστηρίζω αυτό το ε, σημείο. Ich würde gerne drei Anmerkungen machen, möchte aber zunächst dem Kollegen Rübig herzlich Dankeschön sagen für, seinen, für seine gute Stellungnahme.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 Και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Ρούντι, τον εισηγητή και φίλο ε, και να πω πόσο θετικά είναι όλα αυτά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν μπορούν εύκολα να υπερασπιστούν τα συμφέροντα τους. Ε, πρέπει να τονίσω ότι στο κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχουν πολλές ελλείψεις γιατί είναι σημαντικό το θέμα της προστασίας στο διαδίκτυο των δικαιωμάτων των Χριστόν. Υπάρχει το θέμα της ε, πνευματικής ιδιοκτησίας και ουσιαστικά τι μας προτείνεται να δημιουργηθεί ένα παρατηρητήριο ευρωπαϊκό ε, των ε, διαφόρων διοικητικών παραποιήσεων που γίνονται σε θέματα διαδικτύου. Εγώ πιστεύω ότι το κείμενο δεν είναι αρκετά ρωμαλαίο, δεν τα λέει τα πράγματα αρκετά ξεκάθαρα και ίσως στο σημείο 3 πρέπει να, να παρατηρήσω ότι λέγεται η λέξη, να η, έκφραση να, δια, να γίνει η σωστή διαχείριση των εμπορευμάτων μέσω του διαδικτύου. Ε, ε, πρέπει να, να χρησιμοποιήσουμε μια εκφρασή που να λέει ξεκάθαρα να καταπολεμήσουμε τις ε, παραποιήσεις. Ευχαριστώ και δίνω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υποθέτω το ότι ο κύριος Στάντσικα είναι αυτός ο οποίος θα παρέμβει. Ε, διαφορετικά υπάρχει κάποιος άλλος. Ποιος πρόκειται να παρέμβει από την Επιτροπή, δεν υπάρχει κανείς εκπρόσωπος, δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά εφόσον δεν υπάρχει κανείς που θέλει να τοποθετηθεί, θα ρωτήσω τον Ρούμπιχ αν θέλει να πει κάτι ακόμη ή αν θα κλείσουμε το θέμα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω Ε, ε, όσον αφορά αυτά που είπε ο συνάδελφος ο Ντί για τις ε, μικρομεσαίες και δημιουργικές επιχειρήσεις προσπαθούμε να δραστηριοποιηθούμε για το μέλλον και ο καταναλωτής πρέπει να έχει την δυνατότητα ό,τι δημιουργείται και επινοείται να το λαμβάνει στην μητρική του γλώσσα και εφόσον όλη η ομάδα συμφωνεί από αυτού θέλω να την ευχαριστήσω θερμά. Ευχαριστώ. Τελειώσαμε λοιπόν με αυτό το θέμα και αύριο θα γίνει η τελική ψηφοφορία. 10. Ε, έκθεση σχετικά με την ε, πράσινη βίβλο της Επιτροπής για τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο αξιότιμος κύριος Τσίτσεστερ έχει το λόγο και του δίνω τον λόγο και του ε, επιτρέπω να ξεκινήσει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, πάντα ερχόμουν εδώ την κατάλληλη στιγμή και δεν έχανα το χρόνο μου. Θα ήθελα να παρουσιάσω λοιπόν τις τροπολογίες ε, για την έκθεση και θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους κοιόδης εισηγητές μου και τη γραμματεία για την εργασία τους. Ε, πολύ ενδελεχή εργασία στην κατάρτιση διαφόρων τροπολογιών συμβιβασμού. Οπότε έχουμε εδώ μερικά θέματα τα οποία απομένουν απ' έξω ε, μπορούμε να φτάσουμε ίσως να καταλήξουμε σε πραγματική ε, συμφωνία ψηφίζοντας. Εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι τελικά έχουμε φτάσει σε πολύ, καλή, σε πολύ καλές προτάσεις, σε πολύ καλή λύση. Ε, πολλές φορές ε, διαφωνούσα, αλλά θεωρούσα πάντα ότι η Επιτροπή αυτή είναι αρμόδια ε, για θέματα ενεργειακά και ε, το θέμα της ιεράρχησης των αποβλήτων είναι ένα θέμα που πρέπει κανονικά να απασχολεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος πιστεύω και αυτή να το διεκπεραιώνει. Γι' αυτό είχα αυτή τη στάση. Έτσι νομίζω είναι και το σωστότερο. Λοιπόν, δεν θέλω να μακρηγορήσω κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να καλέσω τους συναδέλφους να υποβάλουν σχόλια ή να πούν τι αρνητικό βρίσκουν σε, στις που έχω υποβάλει. Υπάρχουν παράπονα ή παρατηρήσεις, η συνάδελφος Σοφιώνα Χόλ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Τσίτσεστερ για την συνεργασία που μας προσέφερε στους κοιόδης εισηγητές της Επιτροπής πάνω σε αυτή τη γνωμοδότηση και συμφωνώ ότι τελικά καταλήξαμε σε πολύ ε, σωστούς συμβιβασμούς και βοηθητικούς. Επίσης θέλω να πω ότι αυτή η γνωμοδότηση θα πρέπει να επικεντρωθεί στα θέματα της ενέργειας και έχω μια γενικότερη ανησυχία ότι ε, τα ε, βιολογικά απόβλητα δεν έχουν την απαραίτητη προσοχή αυτή που αξίζουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να θέσουμε έναν στόχο ξεκάθαρο για την ε, μεταφορά επίσης των ανανεώσιμων ενεργειών. Και νομίζω ότι το θέμα είναι και το διοικητικό πλαίσιο. Δεν μπορούμε να τα ξεχάσουμε όλα αυτά. Ε, χρειάζεται ε, μια καινούρια οδηγία που να ασχολείται με τα βιολογικά απόβλητα ε, και γι' αυτό θα πρέπει νομίζω να, ε, ότι πρέπει να γίνεται ανακύκλωση σωστά, πρέπει να θεσπιστούν όλα αυτά και έχω καταθέσει μια τροπολογία αριθμός 24 η οποία ασχολείται με αυτό το σημείο. Ε, η Επιτροπή ίσως θα μπορούσε να μας ε, διευκρινίσει τα προβλήματα αυτά ε, για να είναι πιο εύκολα για μας και πέρα από αυτό βεβαίως ευχαριστώ τον κύριο Τσίσεκ για την εργασία του. Ευχαριστώ κύριο Σέντσο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να πω απλώς ότι εκτιμώ ιδιαίτερο αυτό που έκανε ο εισηγητής. Είναι εξαιρετικό το κείμενό του. Όπως είπε όμως και ο ίδιος ο συντάκτης της νομοδότησης, η επεξεργασία βιολογικών αποβλήτων δεν άπτεται μόνο του περιβάλλοντος, ίσα ίσα πιο πολύ έχει να κάνει με τον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας και από προσωπική πείρα μπορώ να σας πω ότι πέραν της ε, ενέργειας η οποία θα μπορούσε να προκύψει από αυτά τα απόβλητα ε, ή των φυτοφαρμάκων που μπορεί να προκύψουν από αυτά τα απόβλητα, η επεξεργασία των βιολογικών αποβλήτων όπως επίσης και η ανάκτηση και ανακύκλωση άλλης μορφής αποβλήτων που είναι απαραίτητα για την ε, πλήρη διαδικασία ανακύκλωσής τους, σημαίνει ότι από το 100% των ε, αποβλήτων ε, μόνο το 50% θα καταλήγει στις κομματερές. Αυτό θα ήταν ιδιαίτερο σημαντικό. Έχω παρουσιάσει και μια σχετική τροπολογία η οποία κάνει μια απόπειρα να πιέσει κάποια κράτη-μέλη όπου δεν γίνεται ε, ανακύκλωση και συγκεκριμένη συλλογή αποβλήτων και εκεί ε, προτείνω να δίνεται μια κάποια αξία σε αυτά τα απόβλητα. Η, το έξοδο θα ήταν ε, ε, ελάχιστο ε, και αν λάβει υπόψη κανείς και τι, ε, τις ζημιές που μπορεί να προκαλέσουν ε, τέτοιας μορφής απόβλητης θα μπορούσαμε ίσως να έχουμε από, κάποιο όφελος και ίσως και κάποιοι θα μπορούσαν να έχουν και κάποιο κέρδος. Και μάλιστα τα κράτη-μέλη θα είναι καθαρότερα και θα έχουν και επιπλέον ενέργεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και δίνω το λόγο στην κυρία Φον Μπρέμ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να συγχαρώ και εγώ με τη σειρά μου τον εισηγητή. Έξοχη η γνωμοδότησή του. Αναπάντοχα καλή. Ε, και μάλιστα ο συντάκτης της νομοδότησης ασχολήθηκε πάρα πολύ και με τις τροπολογίες και με συμβαστικές τροπολογίες που ίσως να μας οδηγήσουν σε αίσιο αποτέλεσμα αύριο. Έχουν ε, κατατεθεί κάποιες συμβαστικές τροπολογίες. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι από αυτού. Ε, υπάρχει η πρώτη συμβαστική ε, τροπολογία, την οποία θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική. Η ανακύκλωση βιολογικών αποβλήτων ε, σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε και πάρα πολύ ε, καλούς ορισμούς, κυρίως όταν μιλάμε για βιοδιασπόμενα απόβλητα. Ε, και επίσης θα πρέπει να δούμε και τι θα γίνει στο μέλλον, διότι στην ιεράρχηση των αποβλήτων είναι σημαντικό να τονίσουμε πόσο σημαντική είναι η επαναχρησιμοποίηση, η δυνατότητα νέας χρήσης, όχι μόνο για την παραγωγή ενέργειας. Η παραγωγή ενέργειας είναι σαφώς σημαντική ε, και για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, αλλά το θέμα του κλίματος δεν πρέπει να το εξετάζουμε μόνο και από την πλευρά της παραγωγής ενέργειας. Θα πρέπει να το εξετάζουμε σε ευρύτερο περιβαλλοντικό πλαίσιο και η χρήση ε, πρώτων υλών μέσω κομποστοποίησης είναι αναπόσπαστο τμήμα όλης αυτής της διαδικασίας. Υπάρχουν ε, οι συμβιβαστικές τροπολογίες οι οποίες ε, θεωρώ ότι ενδυναμώνουν την έκθεση αλλά από πλευράς της ομάδος μου θα ήθελα να τονίσω άλλη μια πτυχή. Θα πρέπει να ε, σταθούμε και σε κάτι ακόμα. Αυξάνεται η σημασία των βιολογικών αποβλήτων, οι δυνατότητες που μας προσφέρονται είναι σημαντικές, επομένως θα πρέπει να υπάρχει και ξεχωριστή οδηγία επί του θέματος. Ευχαριστώ. Ε, ε, Ευχαριστώ πρέπει να ευχαριστήσω τον εισηγητή κύριο Τσίτσεστερ διότι η παρουσίασή του ήταν εξαιρετική και είχε πολύ καλή συνεργασία με όλες τις άλλες σκιώδεις εισηγητές. Δηλαδή προετοιμάσαμε μία σειρά τροπολογιών, είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι για την αυριανή ψηφοφορία και πρέπει να πω ότι θα στηρίξουμε όλες τις συμβιβαστικές τροπολογίες και τις άλλες τροπολογίες, αλλά υπάρχουν υπάρχουν δύο θέματα τα οποία θα ήθελα να τονίσω εδώ. Πιστεύω ότι τα βιολογικά απόβλητα είναι μέρος του μείγματος το οποίο θέλουμε να αντιμετωπίσουμε ε, και ε, αν μιλάμε για βιολογικά καύσιμα δεν πρέπει να παρανοούμε, ε, άλλωστε πρέπει να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε συμβιβαστικές τροπολογίες για να μπορέσουμε να έχουμε μια κοινή αντιμετώπιση. Ευχαριστώ. Δίνω τον λόγο στον κύριο Σπονά. Χρησιμοποίησα το σωστό όνομα για τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με συγχωρείτε αν δεν σας είχα δει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα βεβαίως να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εξαιρετική γνωμοδότησή του. Κατανοώ πλήρως γιατί η Επιτροπή Ενέργειας επικεντρώνεται περισσότερο σε προβλήματα ε, ε των ε, συζητήσεων ε, πάνω στα βιοκαύσιμα, την ενέργεια και το περιβάλλον. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τα μέλη για τις συμβολές τους και ειδικά για τον προλαλήσαντα που μίλησε για την ιεράρχηση πρέπει να θυμούμαστε ότι είναι πάρα πολύ βασικός ο ρόλος της λιπασματοποίησης των αποβλήτων και αυτός είναι ένας τρόπος χρησιμοποίησης της ιεράρχησής τους. Αφεραρχία πρέπει να προβλέπεται κατά κάποιον τρόπο πολύ συγκεκριμένα. Οι αναλύσεις που έχουμε κάνει μας δείχνουν ότι χρειάζεται μια μέθοδος ε, χρησιμοποίησης των ε, αποβλήτων η οποία είναι πολύ πιο χρήσιμη για το περιβάλλον και αυτή είναι η υψηλή ιεράρχηση των αποβλήτων. Υπάρχουν και ορισμένες ε, βεβαίως εξαιρέσεις στον γενικό κανόνα. Αυτό μπορεί να ισχύει για τα βιοκαύσιμα αλλά θα πρέπει να υπόκειται πάντα σε πιο συγκεκριμένη ανάλυση για να διευκρινιστούν όλα τα επίμαχα σημεία. Σε ό,τι αφορά τα, ε, το αίτημα που έγινε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να, να ε, διελευκάνει κάπως το θέμα των βιοκαυσίμων. Ε, νομίζω ότι υπάρχει η αρκετά σαφώς διευκρίνηση μέσα στη σχετική οδηγία. Αλλά η οδηγία αποκλεί την παραγωγή των βιοκαυσίμων μέσα από ανακύκλωση. Αυτό είναι αλήθεια. Και είναι αλήθεια ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης η παραγωγή των βιοκαυσίμων για την ανακύκλωση χρειάζεται ορισμένες νομοθετικές αλλαγές. Επίσης υπάρχουν οι δυνατότητες για τα κράτη-μέλη όταν καταρτίζουν τις εθνικές νομοθεσίες ανακύκλωσης και τους σχετικούς στόχους να δώσουν υψηλότερη αξία στην παραγωγή των βιοκαυσίμων. Νομίζω ότι για την ώρα αυτά είχα να πω κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Μήπως θα ήθελε ο εισηγητής να κάνει ε, συμπληρωματικές παρατηρήσεις. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τα καλά τους λόγια και να επισημάνω δύο σημεία. Το θέμα του ορισμού και της ανακύκλωσης. Εγώ θυμάμαι ότι έγινε μια τεράστια μάχη όταν προσπαθούσαμε να κάνουμε τη διάκριση ε, της ενέργειας για τα απόβλητα ως πηγή μιας ε, νέας μορφής ενέργειας. Ε, Καταλαβαίνω τι λέει η κυρία Χόλς, αλλά εγώ δεν θα είμαι διατεθειμένος να ξαναρχίσω αυτή τη μάχη. Ε, όσο για την ξεχωριστή οδηγία, την οποία εύχεται η κυρία Λαμπέρτη να έχουμε, ξέρετε ότι εγώ είμαι πολύ επιφυλακτικός ε, στην ε, πρόθεση νέων οδηγιών. Δεν είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι είναι αυτό το οποίο πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή. Ε, ας ε, συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε επί του θέματος προς το παρόν. Ολοκληρώνοντας, να πω ότι δέχομαι ότι η γνωμοδότηση είναι κυρίως το θέμα της ιεράρχησης των αποβλήτων και ο τρόπος διαχείρισής τους, ε, αλλά επειδή εμείς δεν είμαστε η Επιτροπή Περιβάλλοντος, θεώρησα ότι ίσως θα πρέπει να σταθούμε περισσότερο στους τομείς που απτούνται τις αρμοδιότητές μας, δηλαδή η ενέργεια για ε, από τα απόβλητα. Ελπίζω να έχουμε ένα καλό έγγραφο, το οποίο θα προκύψει εύχομαι αύριο μετά από την ψηφοφορία και ευχαριστώ τους πάντες για τη συνεργασία τους. Ε, Εγώ ευχαριστώ και έτσι λύεται η συνεδρίαση. Δεν βλέπω να ζητά κανείς άλλο τον ε, λόγο. Άρα ολοκληρώνεται αυτή η, αυτό το σημείο της μερσίας διατάξεως. Τελειώνει η συνεδρίαση για σήμερα και σε πέντε λεπτά θα έχουμε την ε, συνεδρίαση των συντονιστών. Δηλαδή, Δηλαδή θα έπρεπε όλοι οι άλλοι να μπορέσουν να εγκαταλείψουν την αίθουσα για να ξεκινήσουμε. Αύριο θα ξεκινήσουμε στις 9.30 για τις ψηφοφορίες.